Thank you, colleagues. I encourage you to take seat. I would ask those who are leaving not to talk, please, so we can start. Παρακαλώ κάντε λίγη ησυχία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Το έβδομο σημείο της ημερησίας διατάξεως έλεγχος των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εφαρμοστικών μέτρων. Λοιπόν, δίνουμε μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες ελέγχου σε αυτές τις σημαντικές συνιστώσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, όπως τα μέτρα επίπεδου 2. Σήμερα θα εστιαστούμε επί της οδηγίας για υπηρεσίε πληρωμών στην εσωτερική αγορά και κανονισμό για διάφορα τέλη όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Ρία, Όλιβερ Σαλές, ε, Όσον αφορά το PS2, εξεδόθησαν δύο έγγραφα. Έγγραφο συζητήσεως του Δεκεμβρίου του 2015 για το μελλοντικό RTS, για την πιστοποίηση των πελατών και ασφαλή επικοινωνία και το έγγραφο 11 Δεκεμβρίου για το σχέδιο RTS για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών για κοινοποίηση των διαβατηρίων και θα μας ενδιέφερε να ακούσουμε περισσότερα για τα βασικά θέματα και να δώσουμε κάποια συνέχεια όσον αφορά τον κανονισμό για την τέλεια ανταλλαγή στο άρθρο 7 του κανονισμού απαιτεί ότι οι διάφοροι φορείς είναι ανεξάρτητοι όσον αφορά το λογιστικά και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το EBA ξεκίνησε το 8 Δεκεμβρίου δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο RTS, για το διαχωρισμό των πληρωμών μέσω καρτών και η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 8 Μαρτίου και σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τι έγινε με τις διαβουλεύσεις και ποια είναι οι προθέσεις όσον αφορά τα επόμενα ε, βήματα και τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αρία και μετά στους υπόλοιπους για μια σύντομη εισαγωγή. Παρακαλώ να ε, παραμείνετε εντός ε, του ορίου ενός τετάρτου. Ανδρέα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέλη της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω που μου δώσει τη δυνατότητα να ενημερώσω για τη δουλειά που έκανε η ΕΜΠΗ. για το τέλος ε, των συναλλαγών για τις τραπεζικές προμήθειες. Καλωσορίζουμε την εντολή έτσι η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, θα μπορέσει να εποπτεύει καλύτερα την όλη κατάσταση όσον αφορά τις χρηματοστατικές υπηρεσίες, τις λιανικές πληρωμές, επίσης που είναι κάτι πολύ καινοτόμο. Η EBA ε, θέλει να πετύχει τους στόχους του PSD2 και του IFR, να υπάρχει μεγαλύτερο ανταγωνισμός στην αγορά για τις ε, πωλήσει στον τομέα της λιανική. Θα σα δώσω μια αρχική ε, εικόνα για την πρόοδο που πετύχαμε όσον αφορά τι εντολές που ανατέθεσαν. Όπως είπατε, λάβαμε μια εντολή του άρθρου 7,6 6, 6 του IFR όσον αφορά το διαχωρισμό των διαφόρων συστημάτων ε, καρτών πληρωμή και των φορέων ε, επεξεργασία, Έπρεπε να έχουμε τεχνικές προδιαγραφές να θεσπίσουμε όσον αφορά τα σχήματα για τις φυσικές κάρτες και τις φορείς που θα πρέπει να συμμορφώνονται για τα λογιστικά, την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων. Η EBA πληροφορήθηκε ότι αυτή η εντολή εδόθηκε πολύ αργά μετά τι πραγματεύσει όσον αφορά το IFR είχαν λήξει και αμέσω μετά λάβαμε επίγνωση τη εντολή και συγκαλέσαμε ένα εργαστήριο με τη συμμετοχή και από τις δύο πλευρές από... και ξεκίνησε η διαδικασία τον Ιούνιο του 2015. Δημοσιεύσαμε το σχέδιο RTS το Δεκέμβριο του 2015 και κατά τη διάρκεια της περίοδου διαβούλευσης έγινε και μια δημόσια κρόση. Ε, εκεί ε, είχαμε μεγάλη συμμετοχή από 55 ε, άτομα από πάνω από 24 διαφορετικές, ε, διαφορετικούς φορείς. Το σχέδιο RTS αναφέρεται στην ανεξαρτησία την οργανωτική που θα πετύχουμε μέσω λειτουργικού διαχωρισμού, ανεξαρτησία των ανωτέρων στελεχών, αλλά θα προβλέπουμε και κάποιες εξαιρέσει σε συγκεκριμένε περιπτώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει λογιστική ανεξαρτησία, δηλαδή το κόστος θα πρέπει να γίνεται μέσω κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, ABC, και θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και έτσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξασφαλίζει ότι ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων θα μειώνονται. Λάβαμε 16 απαντήσει όσον αφορά τι διαβουλεύσει και τώρα τι αξιολογούμε και θέλουμε να δημοσιεύσουμε το τελικό σχέδιο ε, του RTS τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή εντό του 12 μήνου μετά την έναρξη των εργασιών μα. Θα ήθελα να κλείσω την ενημέρωσή σας για το IFR, γνωστοποιώντας σας ότι ενώ το EBA έχει τη νομική δυνατότητα να αναπτύξει το RTS, παρόλα αυτά δεν έχει εξουσία οποιαδήποτε να εξασφαλίσει ότι το RTS και το IFR εν γέννη θα εφαρμόζονται με συνέπεια από τα χρηματοστατικά ιδρύματα και θα υποπτεύονται από τις εθνικές αρχές. Για να διαδραματίσουμε αυτό το ρόλο, σαν EBA, η νομοθέτηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα έπρεπε να να βάλουν το IFR πλήρως στο πεδίο λειτουργίας της EBA τροποποιώντας ε, τον ιδρυτικό κανονισμό και προσθέτοντας ε, τις, ε, τα διάφορους μηχανισμούς καρτών πληρωμής και τις εποπτικές αρχές στον ορισμό των χρηματοστικών ιδρυμάτων και των αρμοδίων αρχών αντιστοίχως. Ελήψη τέτοια τροπολογία δεν θα πετύχουμε τη σωστή σύγκληση, τόσο ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε στα πλαίσια του κανονισμού του επίπεδου 1. Λοιπόν, έχουμε 11 εντολέ ε, σύμφωνα με το PSD2, 6 τεχνικέ προδιαγραφέ και 5 κατευθυντήριε γραμμέ και έχουμε 12 και 18 και 24 μήνε σαν χρονικά όρια, του ώστε το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την, ε, ε, μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 για το PSD2. Οι εντολέ αφορούν την κοινοποίηση των διαβατηρίων, αδειοδότηση, εποπτεία, αποπτήσει όσον αφορά την ασφάλεια, ε, προ, ε, κοινοποίηση προβλημάτων, δημιουργία ενός μητρώου EBA, δια, ε, διαδικασίες καταγγελιών και ασφάλεια για αποζημιώσεις. Ξεκινήσαμε την επεξεργασία 11, 11 εντολών παράλληλα και ετοιμάσαμε ένα έγγραφο συζητήσεων και ένα έγγραφο διαβούλευση το Δεκέμβριο του 2015, όπως υποθυμίσατε κύριε Πρόεδρε και αυτό πριν το ίδιο το PSD2 ε, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα. Το πιο επίμαχο, η πιο επίμαχη από τις εντολές είναι το RTS όσον αφορά την εξακρίβωση των πελατών και ασφαλή επικοινωνία που αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο βαθμός στον οποίο το PSD2 θα μπορέσει να πετύχει ε, τον στόχο αύξηση ανταγωνισμού εξαρτάται κατά πολύ από το πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο σαν EBA όσον αφορά τερτίας. Δηλαδή πώς οι τράπεζες θα μπορούν να επικοινωνούν με εκείνους που είναι καινούργοι στην αγορά, δηλαδή οι πάροχοι τρίτων, τρίτοι πάροχοι που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς πληρωμών των πρώτων ε, ή να αποκτήσουν πληροφορίες στους λογαριασμούς. Είχαμε 12 μήνες να πετύχουμε το στόχο αυτό που είναι ευαίσθητος και ήδη έχουμε εκδώσει το Δεκέμβριο του 2015 έγγραφο συζητήσεω για μία περίοδο δύο μηνών. Όταν απτύσσαμε αυτά τα RTS, το EBA θα πρέπει να έρθει σε επαφή να, μάλλον να συγκρίνει ε, τα υπέρ και τα κατά. Ένα από τα προβλήματα αφορά την ανάγκη να πετύχουμε μεγάλη ολοκλήρωση στην ενιαία αγορά. Αυτό θα, ε, θα έδειχνε ότι το EBA θα πρέπει να έχει μια ενιαία προδιαγραφή με πολλές λεπτομέρειες εν συγκρίση με τη ζήτηση η διευκόλυνση με την πάρα του χρόνου τη καινοτομία μεταξύ των επιχειρήσεων. Άρα το EBA θα πρέπει να κάνει το αντίθετο, δηλαδή να επιβάλλει απαιτήσει υψηλού επίπεδου που επιτρέπουν σε διάφορε ε, πρότυπα και τεχνολογικέ λύσει να μπορούν να εφαρμοστούν. Η EBA έλαβε 118 απαντήσεις όσον αφορά τη διαβούλευση. Ε, το μεγαλύτερο, δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων ποτέ που δόθηκαν στην EBA στη σύντομη ζωή αυτής. Μόνο η διαβούλευση για την αμοιβή των τραπεζικών υπαλλήλων είχε περισσότερες απαντήσεις. Αυτό μας λέει πολλά Λοιπόν, αξιολογούμε τι απαντήσει και θα εκδώσουμε ένα έγγραφο διαβούλευση στο καλοκαίρι του 2016 και τελικό RTS θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, δηλαδή εντό του 12 μήνου που προβλέπεται από το PSD2. Θα ήθελα να κλείσω γνωστοποιώντα σα ότι είμαστε ικανοποιημένοι πολύ με την επίθεση πρόοδο όσον αφορά τι εντολέ που μα ανατέθησαν. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσουμε σημαντικέ δυσκολίε όμω εκπληρώνοντα τα καθήκοντά μα προχωρώντα λόγω ελλείψεω πόρων. Στον προπολογισμό για το 2016 το EBA δεν έλαβε συμπληρωματικού πόρου για να πετύχει τι εντολέ που ανετέθησαν το καλοκαίρι του 2014. Ζητήθηκε από το EBA να εκτιμήσουμε του αναγκαίου πόρου για να αναπτύξουμε τότε αυτό που προβλεπόταν τέσσερι εντολέ. Ε, τότε είπαμε ότι θα χρειαζόμαστε τρία FTE στο πρώτο έτος, δύο FTE στο δεύτερο έτος και ένα FTE για κάθε χρόνο μετά από αυτό για να αναπτύξουμε τα αναγκαία πλαίσια και να τα συντηρούμε. Όμως ε, δεν λάβαμε κανέναν πόρο και αυξήθηκε ο ρυθμός των εντολών που μας συνετέθη από 4-11 και αυτό μας φαίνει σε μια αρκετά δύσκολη θέση και γι' αυτό δεν μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε όλους τους στόχους εντός των προθεσμιών που μας ετέθησαν και αρχίζουμε να, μειώνουμε, να υποβαθμίζουμε τις προτεραιότητες των τελών, το πρώτο που αφορά τα κεντρικά σημεία επαφής και το άλλο όσον αφορά το μητρό EBA. Ελπίζω ότι αυτή η σύντομη εισαγωγή ήταν επικοδομητή και σας βοηθάει και είμαι πάντα έτοιμος να ακούσω ε, ερωτήσεις μαζί με τον συνάδελφο που είναι υπεύθυνο για προστασία καταναλωτών κλπ. κλπ. Να σας δώσουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημειώνουμε δεόντως αυτά που μας είπατε. Οι ανησυχίε σας είναι και δικές μας ανησυχίες όσον αφορά τους πόρους για την αρχή αυτή, για το EBA. Και λαμβάνουμε υπόψη και αυτό που είπατε για έλλειψη νομικής εξουσιοδότησης ε, για θέματα ελέγχου ε, και την εφαρμογή του IFR. Ο κύριος Σάλες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Να καλημερίζω τα μέλη της Επιτροπής ε, Οικονομικών και σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό θέμα. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Απλά μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι το PSD2 πράγματι θεωρείται ως νομοθεσία ε, σημαντικό ε, νομοθέτημα. Εγκρίθηκε, σας υπενθυμίζω, πέρυσι και βοήθησε πολύ και το Κοινοβούλιο να έχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ανοίγματο ε, των αγορών. Εδώ είμαστε σε ένα πολύ καλό πλαίσιο διαμερισμού ευθυνών από τη μια της ε, Κομισιόν ε, και της CBA της Ένωσης από την άλλη εμείς ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Αφίσμα, εστιάζουμε πλέον ε, στην σωστή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο αυτού του σημαντικού νομοθετήματος ε, και έχουμε γι' αυτό το σκοπό το εργαλείο υποστήριξης των κρατών μελών. Έχουμε εργαστήρια, το ένα έγινε το Φεβρουάριο και το δεύτερο θα λάβει χώρα αύριο. Και θα έχουμε και τέσσερα ακόμη μέσα στο 2016 για τη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο και ίσως περισσότερα του χρόνου, ώστε όλες οι διοικήσεις ε, των κρατών μελών να έχουν την απαιτούμενη γνώση και τα απαιτούμενα εργαλεία στη διάθεσή τους, ώστε να εφαρμόσουν πλήρως ε, την νομοθεσία αυτή μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 που είναι η προθεσμία. Όπως είπε και ο κύριος Αντρέα, υπάρχουν πολλά σημαντικά μέτρα επίπεδου 2 θα πρέπει να εγκριθούν. Θα πρέπει να στεφθεί με επιτυχία αυτή η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Έχουμε εργαλεία, συνεργαζόμαστε, έχουμε τακτικές επαφές, ανταλλαγές, ώστε και νομοθεσία επίπεδου 1 και, και τα μέτρα επίπεδου 2 να καταρτιστούν και να εφαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα σταματήσω εδώ και μπορώ αργότερα να επανέλθω στη συζήτηση αν προκύψει ανάγκη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Βέζεμπεκ. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε να μιλήσουμε για το θέμα. Πρόκειται για τις χρεώσεις για διατραπεζικές ε, συναλλαγές. Ο οργανισμό λοιπόν το 2015 και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο. Η δεύτερη ομάδα κανόνων θα τεθεί ισχύ τον Ιούνιο φέτος. Η είχε μια συνάντηση πλατφόρμα όπως τη λέμε με τα κράτη-μέλη όπου είχαμε τα Υπουργεία Οικονομικών ή και τις εποπτικές αρχές και μιλήσαμε για την εφαρμογή του κανονισμού. Θα έχουμε άλλη μια τέτοια συνάντηση τον Ιούνιο και θα εστιαστούμε συγκεκριμένα στη δεύτερη ομάδα κανόνων. Το βασικό ερώτημα βεβαίω είναι εάν θα λειτουργήσει ο κανονισμό διατραπεζικών χρεώσεων, αν θα έχει τα αποτελέσματα που όλοι θέλουμε. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο μαζί ζήτησαν να κάνουμε μια μελέτη η οποία θα αξιολογεί τα αποτελέσματα του κανονισμού. Έχουμε μια ομάδα ήδη η οποία ασχολείται με το λεγόμενο μηδενικό επίπεδο, δηλαδή ποιε θα είναι οι παράμετροι πριν τεθεί ενισχύ ο κανονισμός για να αξιολογήσουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σήμερα μιλάμε για τις ρυθμιστικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως ήδη υπόθηκε το άρθρο 7 λέει πως τα συστήματα και οι υποδομές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από πλευράς ε, λογιστικής ε, διαδικασίας λήψη αποφάσεων και οργανώσεως και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή αυτή τη στιγμή οριστικοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρατε έχουμε ένα έγγραφο διαβούλευσης ε, δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβρη του 2015, η ακρόαση έγινε το Φεβρουάριο. Γενικώ λοιπόν η Κομισιόν είναι ικανοποιημένη με τη διαδικασία, αλλά ανησυχούμε κάπω για την καθυστέρηση. Είναι λοιπόν σαφέ πω οι προδιαγραφέ δεν μπορούν να εγκριθούν πριν τεθούν ενισχύει οι κανόνε στι 9. Ιουνίου και αυτό σημαίνει πως ε, στον κλάδο θα υπάρχει ένα ερωτηματικό για τις τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθεί ο κλάδος βεβαίως μπορούν να συμμορφωθούν με το σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών όπως δημοσίευσε η EBA αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτές θα είναι οι τελικές μετά οπότε υπάρχει εδώ ένας λόγος ανησυχίας. Έχουμε βεβαίως και ανησυχίες για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Ένα από αυτά είναι πως υπάρχει μια παρέκκληση για την ώρα όσον αφορά τις λεγόμενες καινοτόμες εξελίξεις όπου αμφισβητούμε αν κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ ευρύ. Επίσης υπάρχει η έννοια της εισαγωγής κάποιου επεξεργαστή ε, ο οποίος θα είναι ε, προκαθορισμένος. Αναρωτιόμαστε πως αυτό είναι κάποια διακριτική μεταχείριση. Επίσης αναρωτιόμαστε αν θα υπάρχει κάποιος μηχανισμός για την εσωτερική μεταφορά κερδών για να μην υπάρχει πάλι ακριτική μεταχείριση και ανησυχούμε επίση για το κατά πόσο μπορούν να υποβληθούν αυτέ οι προδιαγραφέ. συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα κώδικα συμπεριφορά για το προσωπικό των εταιριών, αλλά δεν υπάρχουν κυρώσει και δεν ξέρουμε πώ θα εφαρμοστεί στην πράξη. Τέλο, Υπάρχει μία ευρύτατη περιγραφή, μπορούμε να συμφωνήσουμε στις λεγόμενες κοινές υπηρεσίες, αλλά δεν υπάρχουν κριτήρια με τα οποία θα συμμορφωθούν. Οπότε παρακολουθούμε τη διαδικασία και θα ξαναρίξουμε μια ματιά να δούμε αν συμμορφωνόμαστε. Αλλά με ευχαρίστω βεβαίω θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τώρα θα δώσω τον λόγο στους δύο εισηγητές των δύο φακέλων. Παύλος Ολμπαθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές και για την παρουσία τους και για τις εξηγήσει που μας έδωσαν. Με τον κανονισμό ε, ορίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών θα πρέπει να παρουσιάσει ε, τα τεχνικά ρυθμιστικά πρότυπα το Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς έπρεπε να το είχε κάνει. Τελικά υπευλήθη σε διαβούλευση το σχέδιο αυτών των τεχνικών ρυθμιστικών προτύπων 8 Μαρτίου του 2016 ήταν η καταληκτική προθεσμία και από ό,τι κατάλαβα και από τον πρόεδρο της ε, EBA η πρόταση θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2016. Άρα οι επιχειρήσεις θα έχουν ένα μήνα στη διάθεσή τους ε, για να ε, εκπληρώσουν τις ε, προϋποθέσεις. Για να τηρήσουν το άρθρο άρθρου 7 του κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς αντιμετωπίζει αυτή την καθυστέρηση, ποια από... τι έχει να μας πει. Επίσης, θα συστήσει αρμόδιες αρχές αναβολή των κανόνων που θεσπίζονται στο κανονισμό για τις τραπεζικές προμήθειες, ώστε να έχουν περισσότερη, ε, περισσότερο χρόνο οι επιχειρήσεις να τηρήσουν ε, τα όσα προβλέπεται στους κανονισμούς. Πρόεδρος. Ευχαριστώ τώρα ο Αντώνιο Ταγιάννη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της ΕΜΠΑ ε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίασή τους και για τη δουλειά που έκαναν ετοιμάζοντας ε, τη διαδικασία για τις δύο πράξεις για την ε, ταυτοποίηση των τρίτων μερών και για τη ρύθμιση για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών. Είναι καλό να ολοκληρωθεί ένα μέρος της διαδικασίας. Αλλά η όλη διαδικασία είναι ακόμα στην αρχή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΜΠΑ τη βούληση, την πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φαίνεται από την οδηγία που ανακρίθη τον περασμένο Μάιο. Και στις δύο περιπτώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες επικοινωνίας μεταξύ αρχών το Κοινοβούλιο επέμεινε επί μιας ενίας της τεχνολογικής ουδετερότητας των διαδικασιών. Τα πρότυπα και κανόνας δεν θα πρέπει να είναι εργαλεία για να αποκλειστούν φορείς από την αγορά. Αυτό ισχύει και για τις εθνικές αρχές και για τα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτή οι διαδικασίες πρέπει να είναι ενταξιακές, δηλαδή είναι ανοιχτές διαδικασίες, ουδέτερες διαδικασίες. Τεχνική, τρίτα μέρη, καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία. Πρέπει να εμποδίσουμε γραφειοκρατική γλώσσα. Και αφήσει τοποθέτηση να περιορίζει τη συμμετοχή των διαφόρων στο νέο σύστημα που είναι σημαντικότατο που θα πρέπει να καταστήσει πλέον προσβάσιμο το σύστημα πληρωμών που θέλει να στην πρώτη γραμμή να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Θα επαγρυπνεί προσεκτικά το Κοινοβούλιο, θα επαγρυπνά, ούτως ώστε να γίνεται σεβαστή βούλησή του. Το λέω σαφώς, απευθυνόμενος προς την ΕΜΠΑ, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι για μας αντιπροσωπεύει πραγματική προτεραιότητα. αφήσουμε παράμερα, πηγαίνουμε μάλλον από την πλευρά των καταναλωτών και των χριστών Δεν θέλουμε να υπάρχει μια προσέγγιση αποκλεισμού. Αρμοδιότητά μας είναι να επαγρυπνούμε όπως δεν συνέβη αυτό να μην συμβεί. Είμαι σίγουρος από πλευράς ΕΜΠΑ και από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα λείψουν οι θετικές απαντήσεις ε, όσον αφορά αυτές τι εκκλήσεις του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σκιώδης. Όλοι Λουτβίξον έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το θέμα αυτό που συζητούμε, δηλαδή του διαχωρισμού των φορέων πληρωμών και εκείνων που επεξεργάζονται τα στοιχεία και τις πληρωμές. Είναι σημαντικό αυτό για να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Ανταγωνισμός είναι ο σκοπός του όλου κανονισμού. Καλύτερος ανταγωνισμός θα μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις και θα δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά. Δυστυχώς αυτή η συζήτηση παρέμεινε στα επίπεδα νομοθεσίας επίπεδου 2 πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πώς θα εφαρμοστεί η αρχή του διαχωρισμού. Το σχέδιο αυτό των τεχνικών προδιαγραφών είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, ίσως να μπορέσει να λειτουργήσει. Το σημαντικό είναι να μην αποδυναμωθούν οι προσεγγίσεις όσο πλησιάζουμε την τελική εκδοχή. Δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί το κείμενο. Η εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να υλοποιηθεί σωστά. Δεν είναι δεκτό αν σημαντικοί φορείς της αγοράς αρχίζουν να παραβιάζουν τους θεσπιστέντες κανόνες. Για το PSD2 οι εγκριθείς τεχνικές προδιαγραφές είναι αποφασιστική σημασίας για να λειτουργήσει η οδηγία. Χρειαζόμαστε δίκαιο θεμητό ανταγωνισμό ούτω ώστε να λειτουργεί υγιώς και παραγωγικά. Χρειαζόμαστε ισότιμες συνθήκες για τον ανταγωνισμό. Με την νομοθεσία του επίπεδου 1 αυτό γίνεται ξεκάθαρο. Όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ εμπλεκομένων μερών, υπάρχουν διάφορες αρχές που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Πρώτα απ' όλα, απαιτήσει ασφαλείας πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Οι καταναλωτές πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, πάντα ασφαλείς, ανα πάσα στιγμή. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες θα θέσουν εμπόδια για τους παρόντες ε, ε, φορείς που κινούνται στην αγορά και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Θα ήταν απαράδεκτο εάν υπάρχει αποκλεισμό κάποιων φορέων και κάποιων επιχειρηματικών μοντέλων. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα παρόντα μοντέλα για την επεξεργασία των δεδομένων. Είναι αρχή του επίπεδου 1. Πρέπει να γίνεται σεβαστή αυτή η αρχή και για τους κανόνες και τα εργαλεία του επίπεδου 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στις τράπεζες να περιορίζουν την αγορά μέσω λεπτομερών μέτρων Κάτι που ισχύει σαν πρόβλημα σήμερα. Υπάρχει σαν πρόβλημα. Τρίτο, η πάροχη, η, τα τρίτα, η τρίτη πάροχη, τα τρίτα μέρη, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους ε, παραμένουν ελκυστικά για τους καταναλωτές. Δεν θα πρέπει οι τράπεζες να αποφεύγουν τον ανταγωνισμό, υποχρεώνοντας να γίνονται επενδύσεις στα δικά τους συστήματα. Τα τρίτα μέρη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες, υπολογιστές, iPad, κινητά τηλέφωνα. Θα πρέπει να είναι το πλαίσιο όσο πιο ανοιχτό γίνεται στο μέλλον. Όλα αυτά είναι τεχνικά περίπλοκα. Η γενική γραμμή είναι απλούστατη όμως. Πρέπει να δημιουργήσουμε κανόνες που οδηγούν σε ανοιχτό και θεμητό ανταγωνισμό, όπου όλοι οι φορείς της αγοράς έχουν θέση. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τη δέουσα συνέχεια όσον αφορά τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ashley Fox. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω για τον κανονισμό για τα τέλη διατραπεζικών συναλλαγών. Η συνάδελφος για το EBA είπε ότι ενημερώθηκαν αργά για αυτή την εντολή και νομίζω πως είναι και ευγενικός ε, απέναντι στον νομοθέτη γιατί το αίτημα ήρθε στο τέλος του τριμερούς διαλόγου χωρίς καμία διαβούλευση καθόλου με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και είναι λάθος νομίζω να ασκούμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή γιατί άργησε αν επιβάλλουμε ένα τελείως μη ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εξ αρχής και νομίζω πως ως νομοθέτες πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν ζητάμε από την Κομισιόν και άλλες ευρωπαϊκές αρχές να δουλέψουν τελευταία στιγμή και μετά να τους φέρουμε στην Επιτροπή και να τους λέμε «Μα γιατί δεν κινηθήκατε πιο γρήγορα». Η απάντηση είναι ότι αν τους είχαμε δώσει περισσότερο χρόνο και αν δεν το ζητούσαμε στην τελευταία φάση του τριμερούς ε, διαλόγου που ούτως ή άλλως δεν είναι σωστή νομοθετική διαδικασία γιατί εκεί πέρα ε, γίνεται μια σειραφή συμβιβασμών και νομίζω πως το Συμβούλιο και όχι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. Αυτή είναι η απόψή μου λοιπόν για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Τώρα, να ζητήσω και από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή το εξής. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση στις δικές τους κάρτες ε, εις βάρος ε, ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Έχετε λοιπόν ένα παράδειγμα ε, όπου βρήκατε παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού για να επικυρώσουμε αυτό τον διαχωρισμό που προτείνουμε. Και δεύτερον, αν υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις, θεωρείτε πως ένας απλός διαχωρισμός ε, των διαδικασιών λογιστικής και οργάνωσης θα εγγυηθεί ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε φθανές τέτοιες παραβιάσεις. Και αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε να αναφερθώ τώρα στο PSD2, να πω πως στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια ανοιχτή ομάδα εργασίας τραπεζών για να έρθουν μαζί οι τράπεζες και οι εταιρείες ε, χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας ε, για να καταλήξουν σε, ένα, σε μια κοινή προδιαγραφή, τη λεγόμενη API, για να υπάρχει ακριβώς η δυνατότητα διαμερισμού δεδομένων μεταξύ τραπεζών και τρίτων παρόχων. Και έτσι αναφέρεται πως θα είναι ευκολότερο για τις τράπεζες να υπαλληθεύσουν το εάν οι τρίτοι πάροχοι έχουν τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας πριν τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πελατών και έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος απάτης για τους πελάτες. Η ανοιχτή αυτή ομάδα εργασίας μίλησε ακριβώς για τη δημιουργία μιας λευκής λίστας εγκεκριμένων τρίτων μέρων. Μήπως λοιπόν η Κομισιόν θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι παρόμοιο στο πλαίσιο της Ένωσης. Έτσι θα μπορούσαμε ίσως να αντιδράσουμε σε ανησυχίε του τραπεζικού κλάδου, ότι δηλαδή η σωστή ισορροπία μεταξύ ευθύνης ε, και ασφάλειας και του πιεστή 2 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Σόφι Νετφέλντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με την τελευταία πρόταση που έκανε ο Άσλη. Αν δούμε τη δικιά μου τη χώρα, βλέπω πως κάποιες τράπεζες χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή την έλλειψη κοινών προδιαγραφών για να εμποδίσουν νέες εταιρείες να μπουν στην αγορά. Οπότε θα ήταν νομίζω κάτι το ε, θετικό γιατί θα μπορούν τώρα οι τράπεζες να το χρησιμοποιούν για να μειώσουν τον ανταγωνισμό αντί να προετοιμαστούν για το άνοιγμα των αγορών. Εγώ όμως έχω μια διαφορετική ερώτηση γιατί υπήρχε το θέμα της ε, ΣΕΠΑ που ζήτησα της οδηγίας αυτής να περιληφθεί ως ξεχωριστό σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ξέρω ότι δεν το αναφέρατε, αλλά ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς εφαρμόζεται αυτή η οδηγία, γιατί είχαμε μηνύματα από τους ε, πολίτες που έχουν ακόμα προβλήματα και λάβαμε αργά μια ουσιαστική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν δεν το έχει ζητήσει η γραμματεία από την Κομισιόν. Δεν ξέρω, θα έχουμε, θα λάβουμε μια έκθεση τέτοια στο προσοχές μέλλον. Σας ευχαριστώ, δεν βλέπω τον Μακάρθη. Κύριε Ρεϊμόν, ναι παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εκπροσωπώ τον Σβέν Γκίγκολντ και θα ήθελα να κάνω μία δήλωση και τρεις ερωτήσεις όσον αφορά τις πληρωμές πιστοτικών καρτών. Οι πάροχοι πιστοτικών καρτών προσπαθούν να παρακάμψουν την απαγόρευση αυτών των τελών, βάζουν νέες χρεώσεις για τους χρήστες ή αυξάνουν τα τέλη που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό. Κομισιόν έχει δει τέτοιες πρακτικές παράκαμψης ε, του πλαφών ε, στις χρεώσεις. Όπως ορίζει ο κανονισμός και στην περίπτωση που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τι μέτρα θα ληφθούν για να μην παρακάμπτεται το πλαφόν μετά για το pst 2 και την εφαρμογή του πώς ακριβώς θα υπάρξει ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών έτσι ώστε να είναι ασφαλείς ειδικά οι κινητές πληρωμές και αυτές που λαμβάνουν χώρα στον ε, χώρο που γίνεται η πληρωμή. Σας ευχαριστώ. Μάρκο Βάλλη. Δεν έχω παρέμβαση. Θέλω να μιλήσω. Thank you. Ευχαριστώ. Ούτε η Μπάρμπαρα Κάπελ είναι εδώ. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο. Ξανά. Στον κύριο Νρία. Ευχαριστώ για το πρώτο θέμα το οποίο ετέθη για την καθυστέρηση του διαχωρισμού υπό το ε, να πω πως ε, κοιτάξτε είδε οδώς ε, εμείς ε, βεβαίως είμαστε υπέρ του να σεβαστούμε την νομοθεσία και στις περισσότερες περιπτώσεις το κάνουμε αυτό δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε όπως αναφέρθηκε βεβαίως η εντολή ήρθε κάπως αργά στην διάρκεια της διαδικασίας, οπότε γινόταν οι διαπραγματεύσεις ήδη είναι κάτι στο οποίο ακριβώς ζητάμε να μας ενημερώσουν και οι κάρτες ε, και αυτοί οι οποίοι επεξεργάζονται τις ε, πληρωμές. Τώρα το θέμα των πόρων δεν θέλω να το αναφέρω συνέχεια, αλλά πραγματικά βλέπετε πως εδώ πέρα έχουμε την προϊσταμένη και μέχρι πριν από δύο μήνες υπήρχε μόνο ένας ειδικό για τις ε, πληρωμές. Αλλά να τονίσω πως κάποιες, τε, κάποια τέτοια στήματα βεβαίω θα τεθούν ενισχύ μετά την ε, εισαγωγή της νομοθεσίας επίπεδου 1. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Αφορά πάρα πολλές εντολές που έχουν κοινοποιηθεί σε μας. Και κάποια φορά πέρα από την ε, καθυστέρηση τη δικιά μας μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση έγκρισης από την Κομισιόν ή τα δικαιώματα εξέτασης που ασκεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό το οποίο κάναμε λοιπόν για να το αντιμετωπίσουμε είναι πως ξεκαθαρίσαμε, πως ε, αναμένουμε οι τελικές προδιαγραφές να είναι έτοιμες ε, γύρω στη στιγμή στην οποία οι απαιτήσει θα είναι δεσμευτικές πλέον για τις ε, κάρτες και αυτούς οι οποίοι επεξεργάζονται τις πληρωμές. Οπότε θα μπορέσουν να δώσουν μια διαβεβαίωση για την ανεξαρτησία του λογιστικού συστήματος και της επεξεργασίας κτλ. Ήδη αναφερόμενοι σε αυτές τις προδιαγραφές. Και μετά οι αρχές θα μπορούν να τα λάβουν αυτά υπόψη. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε αυτή την μεταβατική ε, περίοδο. Γνωρίζουμε ακριβώς ε, την έμφαση που δίνει το Κοινοβούλιο στην ανάγκη μιας ε, ουδετερότητας των διαδικασιών, ότι δηλαδή οι νέες προδιαγραφές θα είναι ανοιχτές και ότι βεβαίως ε, τελικά θα ωφεληθεί ο τελικός καταναλωτής. Οπότε θα συνεργαστούμε μαζί σας για να ολοκληρωθεί, όπως είπα, το έργο μας. Επίσης με χαρά άκουσα την άποψη ότι οι διάφοροι αρτίες πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Όπως είπα τώρα εξετάζουμε τα σχόλια τα οποία έχουμε λάβει που ελπίζω να οριστικοποιηθούν προσεχώς. Όπως είπα και πάλι δεν προσπαθούμε να εξαναγκάσουμε τις υφιστάμενες εταιρείε σε ένα ενιαίο ε, επιχειρηματικό μοντέλο. Είμαστε υπέρ της αναλογικότητας και να υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές και αρχές ε, όπως απαιτεί η νομοθεσία. Τώρα, δεν ξέρω εάν θέλετε να απαντήσετε, να απαντήσει ο συνάδελφος σε κάποιες ερωτήσει. ερωτήσεις, κάποιες δεν αφορούν εμάς ακριβώς. Πέρα από την δυνατότητα κάποιων ευρωπαϊκών αρχών που θα διασφαλίζουν την πτυχή της ε, ασφαλείας δεν ε, έχουμε εμείς ε, την δυνατότητα να εκπληρώσουμε αυτό τον ρόλο και βεβαίως υπάρχει νομική εντολή για να διασφαλίσουμε μία συνεργασία και σύγκληση μεταξύ των αρχών. Οπότε είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε τη συνεργασία μεταξύ των αρχών όπως υπάρχει σήμερα σε υψηλό επίπεδο. Και θα μείνω σε αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σάλλας. Καταρχάς, σε σχέση με τον κανονισμό της τραπεζικές ε, προμήθειες, πέντε σημεία σημείωσα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για το ερώτημα του κυρίου Θάλμπα κατά πόσον η υλοποίηση του άρθρου 7 πρέπει να αναβληθεί δεδομένης της ε, καθυστέρησης ε, της ε, ΕΜΠ. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο. Οι εθνικές αρχές νομίζω ότι μπορούν να επιβάλλουν τα φόγια αυτής της διάταξης και το άρθρο 7 Εδάφιο 6 λέει ότι μπορεί, δύναται να αναπτύξει πρότυπα, αλλά δεν υποχρεούται προς τούτο. Μπορεί να μην αποφάσισε δηλαδή η ΕΜΠΑ να αναπτύξει πρότυπα. Οπότε και τότε οι εθνικές αρχές θα αναλάμβαναν οι εθνικές αρχές άρα μπορούν να επιβάλλουν την εφαρμογή του άρθρου, μπορούν βέβαια να εξετάσουν ε, το σχέδιο των προτύπων που δημοσίευσε η ΕΜΠΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, αλλά έχουν την διακριτική ευχαίρεια να πράξουν ό,τι θέλουν και δεν νομίζω ότι θα ήταν ευκταίο να αναβληθεί η εφαρμογή. Επίσης, σημειώνω, όσο είπε ο κύριος ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να μετριαστεί ε, ο αντίκτυπο ε, τη εφαρμογή ε, αυτή του κανονισμού και θα δούμε όταν έχουμε και τα τελευταία, μάλλον την τελική εκδοχή των προτύπων με την ΕΜΠΑ, πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Για τον κύριο Φόξ, μακάρι να είχε περισσότερο χρόνο ε, η ΕΜΠΑ, να μα την έδινε δηλαδή και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά όπω σα είπα, δεν ήταν υποχρεωτικό να καταρτιστούν αυτά τα πρότυπα και είναι πολύ καλό που αποφάσισε να εκπώνησε αυτά τα πρότυπα η ΕΜΠΑ και που διαβουλεύτηκε με τον κλάδο, και το ότι υπάρχουν αυτά τα πιο αναλυτικά πρότυπα είναι θετικό. Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν έχουν τη δυνατότητα να τα εξετάσουν. Δεν ήταν όμω κάτι υποχρεωτικό, επαναλαμβάνω. Από αυτήν την έννοια, το αποτέλεσμα είναι θετικό. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει αναβολή και εμείς πιστεύουμε ότι δουλεύει σκληρά, δεν έχουμε κάποια κριτική. Ζητήσατε παραδείγματα αν δηλαδή λόγω του ότι δεν υπήρχε αυτή ο διαχωρισμό ε, προέκυψαν προβλήματα. Ε, εγώ έχω ένα παράδειγμα από τον τομέα τη ενέργεια, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό περιμένετε να ακούσετε. Πρέπει να σα πω ότι τακτικά παίρνουμε ε, τις καταγγελίες ε, των φορέων από την πλευρά τη επεξεργασία που λένε ότι παρέχονται δέσμες υπηρεσιών. Η, η επεξεργασία γίνεται μόνο στο πλαίσιο τη εταιρεία, Αλλά αν δείτε συγκεκριμένα παραδείγματα, Στι κατοχώρε υπάρχει στην περίπτωση, μια περίπτωση τέλος δεκαετίας του 1990 όπου οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να έχουν μια ε, κοινή δομή και αυτό είναι ένα είδος ε, διαχωρισμού. Και οι ίδιες τράπεζες αποφασίζουν στο πλαίσιο του, των καρτών, σε, των πληρώνουμε κάτι ΣΕΠΑ, να έχουν ένα, μια συγκεκριμένη υποδομή την οποία θέτει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που επίσης αναπτύσσει πρότυπα για το διαχωρισμό τέτοιων υποδομών. Τελευταίο σημείο. Εκ μέρους του κύριου Γκίγκολτ μίλησε ένα συνάδελφος για το κατά πόσον οι καταγγελίες για ε, την περίπτωση που δημιουργούνται, που εφευρίσκονται νέα τέλη και προμήθειες. Ναι, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί θα μπορούσε να παρακαμφθεί ο κανονισμός για τις τραπεζικές προμήθειες μόνο αν υπήρχε μεταφορά ε, κονδυλίων. Από αυτόν που τα ζητά σε αυτόν που τα εκδίδει. Δεν σημαίνει δηλαδή κατά ανάγκη ότι έχουμε αυτή την παράκαμψη. Τους ισχυρισμούς τους γνωρίζουμε. Και αν επιληφθούμε, θα το δούμε και με τις εθνικές αποπτικές αρχές που πιστεύουμε ότι είναι και σε καλύτερη θέση ε, να αντιμετωπίσουν πρώτα σε αυτά τα καταγγελίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σάλης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες αντιδράσεις για το στη δύο Βεβαίως συμφωνούμε με τα σχόλια του κυρίου Ταγιάννη και του κυρίου Ρούντιξον. βασική αρχή του PSD2, οι βασικές αρχές που να γίνουν σεβαστές. Ρόλος μας είναι αυτός. Όλες οι αρχικές προθέσεις και τις δύο πλευρές των αριθμιστικών φορέων θα γίνουν σεβαστές. Το κάνουμε αυτό εν μέρη μέσω των προσπαθειών ενσωμάτωσης εθνικό δικαίου, κάτι που κάνουμε που κινούμε τα κράτη-μέλη. Τακτικά παρακολουθούμε αυτή την πορεία. Στα πλαίσια των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καμιά φορά υπάρχουν σχετικές αντιλήψεις ότι οι τράπεζες ή οι παλιοί φορείς αντιστέκονται στους νέους ερχόμενους. Το κατανοούμε. Αληθεύει σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε πολλές επαφές με όλους εμπλεκόμενους φορείς. Καταναλωτές, παρόχους, τράπεζες κλπ. κλπ. Γνωρίζουμε ότι πολλές τράπεζες ετοιμάζονται σοβαρά. Θέλουν να είναι έτοιμες για την πλήρη εφαρμογή του PSD2 προσπαθούν να προβλέψουν τις δέουσες αλλαγές, προσαρμόζονται, προσαρμόζουν τις υποδομές τους, το λογισμικό τους και τον εξοπλισμό τους. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ξέρουμε ότι η αγορά ετοιμάζεται για τις μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν τον Ιανουάριο του 2018. Σύντομα σχόλια. Για προσπάθειες που έγινε στον Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που ο κύριος Φόξ διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το, έργα, το έγγραφο της ομάδας εργασίας για τον ανοιχτό τροπεζικό τομέα. Είμαστε σε επαφές με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, ομάδες προβληματισμού κλπ. Υπάρχει ομάδα προβληματισμού που είναι πολύ δυναμική στον Ηνωμένο Βασίλειο και είμαστε τακτικά σε επαφή. Να υπάρχει κάποια αρχή που θα ελέγχει τους ε, συμμετέχοντες φορείς. Δεν ήταν στο έγγραφο του επίπεδου 1, δεν το πρόβλεψε ο νομοθέτης, δεν το, πρόβλεψε και, δεν το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ινστικτοδός θα έλεγα πρέπει να επικεντρωθούμε στη σωστή εφαρμογή του επίπεδου 1 και τη μασία του ETS και να ακολουθηθούν οι κατευθυντικές γραμμές της ΕΜΠΑ θα το παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς. Η ε, κυρία Εντεφέλτ, η ΣΕΠΑ, το εξετάσαμε ενδελεχώς. Αναβλήθη η προθεσμία από Φεβρουάριο 2014, πήγε στον Αύγουστο του 2014. Έχουμε μείνει δύο χρόνια πίσω όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΕΠΑ. Νομικώς πώς όλα τα κράτη-μέλη έχουν ευθυγραμμιστεί. Υπήρξαν πολλές καταγγελίες πολιτών, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κυρίως με την άμεση χρέωση. Το παρακολουθούμε του σύνεγγις. Ε, προσφύγαμε κατά 10 κρατών μελών. Ε, μάλλον προδικαστικά ή προ, πριν την ε, διαδικασία κατά παράβαση. Σε πιλωτική φάση. Σε τέσσερα κράτη-μέλη, μεγάλα κράτη-μέλη, οι περισσότερες, ε, είχαμε τις περισσότερες καταγγελίες. Μεγάλα κάτι της Ευρωζώνης εννοώ. Και πρόσφατα πρέπει να πω ότι δεν λάβαμε άλλες καταγγελίες από τελικούς χρήστες. Έχουμε την εντύπωση ότι οι περισσότερες αρχές κατέβαλαν προσπάθειες το τελευταίο δεκάμινο, εξασφαλίζοντας ότι μας κοινοποιούν για την αρμόδια αρχή που θα ασχοληθεί με το θέμα. Με τα χαρά να δώσω και άλλε πληροφορίε. Δημερό αν απαιτείται κάτι τέτοιο. Και ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. που δόθηκε στην ερώτηση της συναδέλφου Ιντβελτ. Ελπίζω να είναι ικανοποιημένη από την απάντηση. Λοιπόν, τελειώνουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τον Αντρέα Ρία τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σημαντική αυτή ανταλλαγή απόψεων επί σημαντικής συνιστώσας της ενίας αγοράς και της χρηματοπιστωτικής ολοκληρώσεως διακοπή θα τα ξαναπούμε στις 11 και 45 με τις ψηφοφορίες.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Για να ψηφίσουμε. Α κάνουμε μια δοκιμή. Ξεκινά λοιπόν η δοκιμή μας. Να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν δουλεύει το σύστημα. Να ψηφίσετε όλοι έτσι για τη δοκιμή. Έξοχα. Εντάξει, υιοθετείτε το, η δοκιμή και το κείμενο. Πρώτη έκθεση. Ντάριος Ροζάτη. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, Τροπολογία 81 υπέρ κατά α, έλεγχος για την 81 άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά έλεγχος για την 84 άρχεται πέρας απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω χέρια έλεγχος λοιπόν λέω ότι απορρίπτεται ας ελέγξουμε Πέρας. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 88. Άρχεται. Πέρας απορρίπτεται τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές έλεγχος νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά σε ελέγξουμε ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω από ό,τι πρέπει. Καλώς πέρας. απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τοπολογία 96 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 96 άρχεται πέρας απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά 97 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 97 άρχεται. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 98. Πέρας εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά γίνει έλεγχος άρχεται πέρας απορρίπτεται με μια ψηφοδιαφορά τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος πέρας Α, απορρίπτεται συγγνώμη έκανα λάθος 108 υπέρ κατά έλεγχος Rejected. Απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά έλεγχος για την 110 Πέρας. Απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνω τον έλεγχο το EFTD να σηκώνει το χέρι διαφορετικά πρέπει να κάνω έλεγχο κάθε φορά κάνουμε έλεγχο Πέρας. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 113 άρχεται. πέρας απορρίπτεται 114 υπέρ κατά άποχες ίδια διαφορά αλλά σε ελέγξουμε δεν βλέπω τα χέρια σας πέρας απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά έλεγχος πέρας απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ α όχι τροπολογία 6 τα συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 122 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 125 πέρας απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά έλεγχος για την 128. Πέρας. Απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. πέρας απορρίπτεται 130 είπε. κατά άποχες απορρίπτεται έλεγχος άρχεται πέρας απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά έλεγχος για την 137 άρχεται Πέρασε. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Μέσω ισοψηφίας. 139 υπέρ. Κατά έλεγχος άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται. εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 141 πέρας ισοψηφία απορρίπτονται 142 υπέρ κατά έλεγχος Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για τη 15. Ξεκινάει. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η διαφορά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 34 υπέρ κατά έλεγχος πέρας απορρίπτεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 37 Α, 37 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχους Πέρας απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά έλεγχος για τη 42 ξεκινάει. Πέρας. Απορρίπτεται. Μια Μία ψήφος διαφορά. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά έλεγχος ξεκινάει. Ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο πέρας απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ήδη 47 άρχεται. Αγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Δύο συνάδελφοι που δεν ψήφισαν ακόμα. Πέρας. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το έλκτη είναι υπέρ ή κατά. Α, δεν σας είδα. Έλεγχος λοιπόν. Πέρας. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. αποχές έλεγχος να σηκώνετε το χέρι ψηλά πέρας απορρίπτεται 64 είπε, κατά έλεγχος για την 64 έρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά 65 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, 65 άρχεται η σουφορία. Πέρας. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 66. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 69 υπέρ. Κατά. Έλεγχος της 69 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Yeah, quicker query uh, directly we would. Vote is closed. Πέρας. Rejected. Απορρίπτεται. Τρία. Δεν ψηφίζουμε. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 72 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 73 είπε. Κατά. Έλεγχος για την 73. Πέρας. Εγκρίνεται. 74 είπε. Κατά. Ήδη διαφορά. Εγκρίνεται 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 και 68 ξεχωριστική και οι δύο μονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική. 67 και 68. Άρχεται. Vote is closed. Πέρασε. Απορρίπτεται. 68 το ίδιο ονομαστική ψηφοφορία, η διαδικασία. Secretariat is telling not... Η γραμματεία λέει ότι δεν είναι ταυτόσιμες και πρέπει να ψηφιστούν και οι δύο. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη δεύτερη. Άλλος ένας που πρέπει να ψηφίσει. Πέρας. Απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται Πέρασε. απορρίπτεται 39 υπέρ όχι λέει ο πρόεδρος καταπίπτει 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος 135 άρχεται πέρας απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε το τροποποιηθέν κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία που Πέρας. 46 υπέρ. 0 κατά 11 αποχές. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. One too many. Ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Okay, but is closed. Πέρας. 45 ψήφοι υπέρ, 0 ψηφι εναντίον, 11 αποχές. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάμε τώρα παρακάτω. draft report... Uh, Σχέδιο εκθέσεως Γιάχο Φαντσέκερ με σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα νομίσματα. Λοιπόν, συμβαστική Α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ινκο 9. Ινκο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Γ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά υπέρ υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να την επαληθεύσουμε έρχεται η ψηφοφορία ενδιαφέρον πολιτικός συνδυασμός πέρας λοιπόν εγκρίνεται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 αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές 85 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική H μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται η συμφορία. πέρας ναι απορρίπτεται συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, αιτιολογική σκέψη ένα. μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί νομίζω ε? ναι ωραία αλλά βεβαίως τροπολογία 3 να τις ψηφίσουμε όλες ωραία υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε τη 13 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε άρχεται ψηφοφορία ονομαστική ψηφοφορία Vote is closed. Πέρασε. 54 υπέρ, μία κατά 2 αποχές. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα ψηφίζουμε την έκθεση Στόλογιαν με τον μακροσκελέστερο τίτλο που έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής οπότε δεν θα τον διαβάσω Δουπουχουά, Έσοχα και Σέδεσου Λοιπόν, συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική Β υπέρ με προφορική τροπολογία των πρασίνων υπέρ κατά Να την επαληθεύσουμε. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ. Κατά υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 με προφορική τροπολογία δεκτή ναι, υπέρ με συγχωρείτε. Κατά. Να την επαληθεύσουμε, κύριε ψηφοφορία. Πέρασε. Τεκτή. 52 υπέρ. Κατά. να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική δέλτα, μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά. Να την επαληθεύσουμε άρχη τη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 11 της κοντ με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 66 υπέρ κατά άρχεται ψηφοφορία 66. Πέρας. απορρίπτεται. Συμβαστική AIDS. Υπέρ. Με μέρος όχι. Με προφορική τροπολογία, με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε λοιπόν. Άρχιε ψηφοφορία. Με την προφορική τροπολογία. Η συμβαστική με την προφορική τροπολογία. Δεν έχουν ψηφίσει όλοι οι συνάδελφοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την αρχική AIDS λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτή. 71 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική Α, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 10 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική J α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 87 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μια ψήφο διαφορά. 88 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 89 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε και αυτήν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, απορρίπτεται με μια ψήφο διαφορά. 90 με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο όχι λοιπόν συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ν με την προφορική τροπολογία και χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται μπορούμε όμως να την επαληθεύσουμε μέρος πρώτο με προφορική τροπολογία πέρας ναι απορρίπτεται μέρος δεύτερο δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το πρώτο. Μέρος δεύτερο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Υπέρ του δεύτερου μέρους. Υπέρ. Κατά. Να παλιτεύσουμε το δεύτερο μέρος. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Μέρος τρίτο. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μέρος τέταρτο. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 99 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Συμβαστική όμικρον υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 18 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Αιτιολογική σκέψη 1 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχέ δεκτό. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχέ δεκτό. Τροπολογία 2 υπέρ, αιτιολογική σκέψη 2 υπέρ, κατά αποχέ δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχέ δεκτή. Αιτιολογική σκέψη 3 υπέρ, κατά αποχέ δεκτή. Αιτιολογική σκέψη 3 α με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τη λογική σκέψη 4 11 αρχικό κείμενο υπέρ κατά ε, δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αρχικό κείμενο 13 και 14 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Αρχικό κείμενο της 15 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 15 β προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτό. Αρχικό κείμενο 16 και 18 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 21 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τι, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τι, A, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική UA υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική V υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. τεολογική σκέψη J, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ετολική σκέψη M. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 52 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, μάλλον πέντε αποχές, συγγνώμη, καμία ψήφος κατά. Πάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, Τρεμόσα η Μπαλθέλης για την παρακολούθηση εφαρμογής του νοσιακού δικαίου ετήσια έκθεση 2014 είναι η τελευταία ψηφοφορία για σήμερα συμβιβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική A ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβεβαστική BA. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεβαστική C. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E δύο τμήματα έχουμε. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Παρακαλώ. Φαίνεται να είναι το EFTD πέρα, αλλά τέλος πάντων. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F, υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38, υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 39. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Ελέγχουμε την 63. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. και η συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται έλα συμβιβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78, υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε την 71, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Την 78, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα, ψηφίζουμε το κείμενο συνολικά όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 24 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την συνεδρίαση, επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα το μεσημέρι. 23 Μαΐου Δευτέρα. 3 με 6.30. Και τρίτη, 9 με 12.30. Πέρα συνεδρία σας. Ευχαριστώ.